αναφέροντας ή ε, επιτυγχάνοντας και την ε, συνένεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα τα πούμε εν το χρόνο. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Υπουργό, την κυρία Κρέιτον. Έτσι λοιπόν ε, ολοκληρώθηκε η συζήτηση και ως επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης Έχουμε ένα θέμα που έχει προτείνει η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων. Είναι μια προφορική ερώτηση προ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματο τη Στοχόλμη και τη θέσπιση του χώρου ελευθερία, ασφάλεια και δικαιοσύνη. Ε, θα ξεκινήσουν ε, καταρχήν οι συντάκτε αυτή τη ερώτηση, ο κύριο Μπέρλιγκουερ, για τρία λεπτά. Signor Presidente, Το e, πρόγραμμα <clears throat> di Stoccolma adottato 2010 το 2010 η Επιτροπή υπέβαλε ένα σχέδιο δράσης ε, σχετικά με μία σειρά από που πρέπει να επιτευχθούν μέχρι το 2014. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έλαβε δύο φορές ε, σημαντικές αποφάσεις το 2009 και αργότερα το 2010. Κατόπιν λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε ένα πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση αυτού του προγράμματος δράσης της Στοκχόλμης. Τώρα αυτό το πρόγραμμα έχει φτάσει στη μέση της διάρκειας ζωής του. Η Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, των Πολιτικών Ελευθεριών και ε, των σταγματικών Υποθέσεων, αυτές οι επιτροπές αποφάσισαν να αξιολογήσουν την μέχρι τώρα πρόοδο για να δουν τι πρέπει να γίνει περαιτέρω. Και εγώ προτείνω ένα πράγμα ή κάνω μια ερώτηση και στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή που είναι η εξή. Υποβάλαμε αυτή την ε, προφορική ερώτηση με στόχο να εστιάσουμε την προσοχή μας στη συγκεκριμένη εφαρμογή των ε, ευρωπαϊκών διατάξεων. Όλα αυτά λοιπόν τα χρόνια έχουμε μπορέσει να ε, συγκεντρώσουμε ένα κόρπους γιούρις, ευρωπαϊκό κόρπους γιούρις, το οποίο οδηγεί στην ε, ολοκλήρωση των ε, δικαιωμάτων και στην ενσωμάτωσή τους σε αυτό. Καλούμεθα λοιπόν να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα και αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι απαριθμούμε τις διατάξεις που έχουμε γκρίνει, δηλαδή τις ε, διατάξεις που έχουν συμπεριληφθεί σε νόμους ή σε άλλες νομοθετικές πράξεις. Εκείνο που έχει σημασία είναι οι πολίτες. Τι φτάνει στους πολίτες σχετικά με αυτές τις ε, τελευταίες εξελίξεις. Ε, γιατί τελικά μόνο ένα μικρό κομμάτι φτάνει στους πολίτες και αυτό προκαλεί τον κίνδυνο να ματαιωθεί το έργο μας. Γιατί τελικά εμείς από ό,τι φαίνεται καταβάλουμε πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια από αυτήν που βρίσκει απήχηση στην ευρωπαϊκή κοινωνία. Επιθυμούμε λοιπόν στην αξιολόγηση ε, αυτής της ε, ενδιάμεσης έκθεσης, να ακούσουμε την άποψη του Συμβουλίου ε, πώς ακριβώς έφτασαν σε αυτό το αποτέλεσμα μέχρι σήμερα και τι πιστεύουν ότι συμβαίνει στην πράξη. Γνωρίζουμε λοιπόν το τι έχει υιοθετηθεί και πρέπει να δούμε τι μπορεί να υιοθετηθεί ακόμα. Διότι ο νομοθέτης ε, έχει ως αντικείμενο να εκπονεί διατάξεις. Όμως ο κυβερνών έχει κατά κύριο λόγο μέλημα να επιτυγχάνει αποτέλεσμα από αυτές τις διατάξεις κυρίως στην Ευρώπη όπου είμαστε όλοι νομοθέτες ακόμα και η εκτελεστική εξουσία έχει το μονοπόλιο της νομοθετικής πρωτοβουλίας Άρα δηλαδή με τον τρόπο αυτό ε, μπορεί να υπονομευτεί η αποτελεσματικότητα του ε, νομοθετικού σώματος. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θέλουμε να έχουμε συγκεκριμένα στοιχεία και θέλουμε να ενημερωθούμε καλύτερα γιατί καταρτήσαμε αυτό το πρόγραμμα της Στοχόλμης και θέλουμε να ξέρουμε τι ακριβώς αποτελέσματα έχει επιφέρει. Ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρο. Ε, ευχαριστούμε τον κύριο Μπελιγκόρ. Ο κύριο Λόπε Αγκουιλάρ για τρία λεπτά, παρακαλώ. Το 2009 το Δεκέμβριο εκρήθηκε αυτό το πρόγραμμα με στόχο να αξιολογήσει ε, στα μέσα της θητείας ε, την εφαρμογή. Τώρα έχουμε περάσει κατά πολύ τη μισή θητεία και είναι ένα θέμα ηθικό. Ε, και είναι δύο τα πράγματα που μας απασχολούν. Πρώτο, ποια ήταν τα αποτελέσματα μέχρι σήμερα του προγράμματος και το δεύτερο ερώτημα, ποια είναι τα βασικά στοιχεία που θα μπορούσαν να εμπνεύσουν το πρόγραμμα που θα διαδεχθεί το πενταετές της Οχόλμης, δηλαδή το 2014-2019. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ένας χώρος ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης, βεβαίως. Αλλά θα πρέπει να δούμε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Έχουμε δει προόδους χωρίς καμιά αμφιβολία ε, στην ποινική ε, δικονομία και στα δικαιώματα ε, όσων διώκονται ή κατηγορούνται, αλλά απέχουμε πόρο από την ολοκλήρωση για να κυρωθεί η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Έχουμε δει ένα δίλημα στην Κοπεχάγη Ξέρουμε ποια είναι τα κριτήρια της Κοπεχάγης. Διάκριση των εξουσιών, δημοκρατία για την προσχώρηση, για να μπει κανεί να γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή είναι μέλος όμως. Πού είναι οι εγγυήσει, οι δικονομικέ, η πρόσβαση σε έγγραφα ή διαφάνεια. Αυτή τη στιγμή συζητούμε ένα φιλόδοξο πακέτο, μια δέσμη για την προστασία, ε, οδηγία και κανονισμό που επίσης πόρο απέχει από την ολοκλήρωση. Έχουμε δει ε, προκλήσεις και οπισθοδρόμηση στην ελεύθερη κυκλοφορία των προσώπων ε, από διάφορες κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλουν να ξαναυψώσουν σύνορα μεταξύ των κρατών μελών. Μα ε, εκεί που θεωρούν οι πολίτες την ελεύθερη κυκλοφορία από τα μείζωνα επιτεύγματα της ίδιας της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της ιστορίας της, όχι μόνο του χώρου ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης. Θα πρέπει καλύτερα να προστατεύουμε τους ευρωπαίους πολίτες Υπάρχουν μεγάλες προκλήσεις και εκκρεμίες και είδαμε να αναδύεται με πάρα πολύ σφοδρότητα μια κρίση που δεν είναι μόνο οικονομική και νομισματική αλλά και πολιτική και νομιμότητας δημοκρατικής αλλά και ηγεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν εκτοξευθεί οι λαϊκισμοί και αυτό συνιστά ομή πρόκληση στα θεμέλια και στις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι μέλη γενέστε λοιπόν με το πρόγραμμα της Στοχόλμης, τι μπορούμε να κάνουμε για να εμπνεύσουμε το επόμενο πενταετές πρόγραμμα υπήρχε προηγουμένως το πρόγραμμα της Χάγης και πριν από αυτό του Τάμπερε. Μετά τη Στοχόλμη λοιπόν, τι θα είναι το πρόγραμμα αυτό για να μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο όπως ορίζει η συνθήκη της Αβώνας. Τρία χρόνια μετά τη θέση σε ισχύ τη και τρία χρόνια μετά την έγκριση του προγράμματος της Στοχόλμης θα πρέπει οπωσδήποτε να δώσουμε απαντήσεις για μεγαλύτερη ασφάλεια των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών στην Ένωση ακόμα και σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εξαιρεί ε, στην ποινική δικαιοσύνη τη συνεργασία των διοκτικών και αστυνομικών αρχών. Αυτό θέλουμε να μάθουμε την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να απαντήσουμε στις τρεις ερωτήσεις της προφορικής ερώτησης. Διακυβεύεται η αξιοπιστία του ευρωπαϊκού εγχειρήματο, η εμπιστοσύνη των πολιτών στο εγχείρημα αυτό και πιστεύουμε ότι αυτή είναι η τελευταία η εσχάτη ευκαιρία που έχουμε για να δώσουμε μια απάντηση στα δικαιώματα των πολιτών που είναι ο λόγος ύπαρξης της Ευρώπης. Αν δεν το κάνουμε τώρα, ε, πιθανώς να είναι πολύ αργά όταν θα προσπαθήσουμε στην επόμενη θητεία. Ευχαριστώ πολύ κύριε Λόπες Αγγελά Και τώρα ο συνάδελφος Κασίνη για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πρόεδρε και εγώ διερωτώ με ε, ποιο είναι το νόημα αυτής της ε, ερώτησής μας. Ε, έχει υπάρξει έκθεση πρωτοβουλίας των τριών επιτροπών που συνέταξαν αυτήν την ε, προφορική ερώτηση. Υπάρχει και το άρθρο 51 και οι επιτροπές ε, λοιπόν έχουν αναφερθεί στο ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Τότε δηλαδή δεν είχε ακόμα τεθεί σε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνας. Τότε πρόκειται για μια πρώτη εφαρμογή του άρθρου 51. Ε, πρόκειται για την συμμετοχή τριών επιτροπών και αυτό καταδείκνυε το πόσο σημαντικό ήταν το θέμα. Το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης αφορά το σύνολο του τρίτου πυλώνα του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, το οποίο εισήγαγε η συνθήκη της ε, Λισαβόνας. Στόχος είναι να υπάρχει η κυριαρχία, ε, η ανεξαρτησία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για θέματα που είναι σημαντικά για τους ευρωπαϊκούς λαούς, έχουν σχέση με την ελευθερία και την ασφάλεια. Ο ενιαίος ευρωπαϊκός χώρος είναι ε, καθοριστικής σημασίας και αυτό αναφέρεται και στη συνθήκη του Άμστερνταμ. Ε, πρέπει λοιπόν να δώσουμε εντολή στην Επιτροπή να μας ενημερώσει σχετικά με την πρόοδο με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Τώρα όμως ε, αυτό το έχουμε πράξει και παλαιότερα στις 25 Νοεμβρίου ε, ρωτάμε, την Επιτροπή τι ακριβώς έχει υλοποιηθεί και τι υπολείπεται ακόμα, ποιες είναι οι δυσκολίες ε, και τι μπορεί να γίνει για να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες αυτές. Ε, επίκυνται οι εκλογές του 2014, θα υλοποιηθούν σε μια περίοδο κρίσης, όχι μόνο οικονομικής αλλά και εμπιστοσύνη απέναντι προς την Ευρώπη. Η συμμετοχή των λαών μειώνεται όλο και περισσότερο στις περισσότερες χώρες, ακόμα και σε εκείνες που ίδρυσαν την Ευρώπη, που την εμπλούτησαν, ακόμα και σε αυτή τη χώρα που είχαμε την κατάρρευση του τείχους του Βερολίνου. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε. Παρά την κρίση ε, και τις εκλογές που θα γίνουν σε περίοδο κρίσης, πρέπει να υπάρξει κάποια ανάκαμψη σε αυτό το πρόγραμμα ε, Μέχρι τις τελευταίες εκλογές ε, οι συζητήσεις ε, ήταν γύρω από την εσωτερική πολιτική. Ε, πρόκειτο για ένα είδος ελέγχου των κυβερνήσεων. Τώρα όμως τίθεται και το ερώτημα ναι ή όχι στην Ευρώπη. Πρέπει να δείξουμε με αποτελεσματικό τρόπο στους πολίτες το ότι έχουμε επιτύχει, ελευθερία, δικαιοσύνη. Αυτά είναι σημαντικά αγαθά και γι' αυτό πρέπει να δώσουμε συγκεκριμένες και πιστικές πληροφορίες. Ε, θα μου επιτρέψετε να υποβάλω τρεις συγκεκριμένες ερωτήσεις. Η πρώτη είναι τα νέα αυτά μέσα με ποιο τρόπο έχουν επηρεάσει ε, την διεκδίκηση των στόχων που αναφέρονται στη, στο πρόγραμμα Στοχόλμης. Δεύτερον, Επιτροπή με ποιο τρόπο προτίθεται να επιτύχει καλύτερη εμπιστοσύνη από πλευρά πολιτών ε, για να είναι ε, πιο ουσιαστικά τα ερωτήματα των πολιτών και τρίτον ε, τι προτίθεται να κάνει η Επιτροπή σχετικά με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ευχαριστούμε πολύ. Εκ μέρου του Συμβουλίου η κυρία Κρέιτον, η Υπουργός κυρία Κρέιτον. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ευκαιρία να αξιολογήσουμε την πρόοδο στο πρόγραμμα τη Στοχόλμη. Το ζήτημα είναι τεράστιο, δεν έχουμε αρκετό χρόνο. Αναγκαστικώ θα περιοριστώ σε μια σύντομη απάντηση. Σίγουρα έχει σημειωθεί πρόοδος, θα συνεχίσουμε στον δρόμο αυτό, στον τομέα. Το Συμβουλίο Δικαιοσύνη και Ιστορικών Υποθέσεων τον Ιούλιο προέβη σε ενδιάμεση αξιολόγηση του προγράμματο τη Στοχόλμη. Η συζήτηση μεταξύ των Υπουργών επικεντρώθηκε στην κατάσταση υπό Κυπριακή Προεδρία. Η επισκόπηση περιείχε αξιολόγηση τη πρώτου όλου του τομεί, άσυλο και μετανάστευση, αστικέ υποθέσει, εσωτερική ασφάλεια, προστασία του πολίτη και εξωτερικέ σχέσεις στον τομέα της δικαιοσύνης και των ιστορικών υποθέσεων κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου η Κυπριακή Προεδρία ενημέρωσε τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου γραπτός για το αποτέλεσμα της συζήτησης στο Συμβουλίο. Σημείωνε συγκεκριμένα και παραθέτω ότι η συζήτηση στο Συμβούλιο κατέληξε σε γενική ικανοποίηση στον αφορά την πρόοδο, επιβέωσε την βούληση του Συμβουλίου να προωθήσει περαιτέρω το πρόγραμμα της Στοκχόλμης, ώστε να δημιουργηθεί πραγματικά ένας χώρος για πολίτες ελευθερίας, ασφαλής και δικαιοσύνης. Η χρησιμότητα του προγράμματος που γραμμίστηκε από διάφορες αντιπροσωπίες, πρόκειται για ένα μέσο υλοποίηση διαφόρων προτεραιοτήτων. Οι Υπουργοί επαναβεβαίωσαν την προσήλωσή τους στους τρεις αυτούς πυλώνες και στην προστασία των ατομικών δικαιωμάτων. Δεν θα σας δώσω εξαντλητικό κατάλογο των μέτρων που συνομολογήθηκαν το 2010, όμως θα ήθελα να τονίσω μερικά από αυτά. Στον τομέα του ασύλου και της μετανάστευσης θεσπίστηκαν ολοκληρωμένα μέτρα για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου. Έχουμε πια καταλήξει ως προς το θέμα, είμαστε, ή τουλάχιστον είμαστε πολύ κοντά. Επίσης το πρόγραμμα πανεγκατάστασης και η οδηγία για του υπηκόου τρίτων χωρών και το δικαίωμά να διαμένουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσον αφορά τα επιχειρησιακά μέτρα, έχουμε το σύστημα θεωρήσεων, το VIS, το σύστημα πληροφοριών Schengen 2 είναι πλέον επιχειρησιακά έτοιμο από τον περασμένο Απρίλιο. Στο μέρο τη δικαιοσύνη είχαμε την οδηγία για τι ελάχιστε προδιαγραφέ, ελάχιστε απαιτήσει για την υποστήριξη των θυμάτων εγκληματικών ενεργειών και επίση τον κανονισμό για την αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασία σε αστικέ υποθέσει. Όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια και τα σχετικά μέτρα, σημαντικός αριθμός ε, σημαντικών οδηγιών υπερψηφίστηκαν για την καλύτερη προστασία από επιθέσεις στον κυβέρνοχώρο, πρόληψη της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών στο διαδίκτυο, βελτίωση προστασίας των παιδιών που είναι θύματα τέτοιων ενεργειών, οδηγία για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εμπορίου ανθρώπων. Το Συμβουλίο εν γέννη έχει την άποψη ότι τώρα πρέπει να εστιάσουμε την προσοχή μας στην εφαρμογή της ήδη θεσπιστής νομοθεσίας και να βεβαιωθούμε ότι τα θεσπισμένα μέτρα είναι πλήρως λειτουργικά. Όσον αφορά τις θεσμικές προσαρμογές, το Συμβούλιο πιστεύει ότι η νομοθετική διαδικασία αποδίδει και τα δύο νομοθετικά όργανα συνεργάζονται ικανοποιητικά στον τομέα Τη δικαιοσύνη και των ιστορικών υποθέσεων. Έχουμε ένα λειτουργικό πλαίσιο πλέον. Οι διατάξει τη Λισαβόνα ήδη έχουν αποδείξει τη χρησιμότητά του. Έχουμε μια μόνιμη επιτροπή στο Συμβούλιο που διασφαλίζει την λειτουργική συνεργασία στον τομέα τη εσωτερική ασφάλεια με μέτρα όπω η ρήτρα αλληλεγγύη, η οποία στο μέλλον δεν υπάρχει καμία αμφιβολία θα μα βοηθήσει να ενισχύσουμε περαιτέρω την μεταξύ μας εργασία. Η δημιουργία επίσης της υπηρεσίας εξωτερικής δράσης συμβάλλει και αυτή στον καλύτερο συντονισμό τόσο της εξωτερικής όσο και της εσωτερικής διάστασης. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι βουλευτές, είμαστε αρκετά ικανοποιημένοι όσο αφορά την πρόοδο που σημειώσαμε. Φυσικά δεν πρόκειται να επανεπαυθούμε. Και αυτό δεν το λέω μόνο εξ του Συμβουλίου αλλά και του Κοινοβουλίου. Τα θεσμικά όργανα πρέπει να αποδείξουν στην πράξη πλέον την προσήλωσή μα στην προσπάθεια επίτευξη πρόοδου στο πρόγραμμα τη Στοκχόλμη με στόχο τη δημιουργία χώρου ενό ανοιχτού χώρου ελευθερία, ασφαλεία και δικαιοσύνη στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ, κύριε Κρέιτσον. Ο Επίτροπος κ. Σπόρτσα έχει το λόγο. Since the speak a Latin language, Δεδομένου ότι άκουσα λατινογενείς γλώσσες από τους ερωτώντες, επιτρέψτε μου να ξεκινήσουμε τα τελικά. Ευχαριστώ λοιπόν τους ερωτώντες για αυτή την ερώτηση που έθεσαν και διότι ζήτησαν από την Επιτροπή όχι μόνο τον κατάλογο όλων εκείνων που επιτεύχθηκαν κατά τη διάρκεια εφαρμογή του προγράμματος της Στοχόλμης, αλλά θέλω να ενημερωθούν και για τα εμπόδια που προέκυψαν κατά την εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Επίσης, θέλω να σας πω ότι έλαβα ιδιαίτερα υπόψη με αυτά που είπε ο κύριος Μπερλιγκουέρ που είπε ότι εντάξει καλό είναι να υπάρχει ένας κατάλογος αλλά σε τελική ανάλυση τι εφαρμόστηκε από αυτό το κατάλογο και αυτό το πρόγραμμα. Σε μια χώρα που γνωρίζω πάρα πολύ καλά, στη Μάλτα, η Μάλτα το 2007 εισήχθη στο σύστημα Schengen. Σήμερα λοιπόν είναι δυνατόν να οδηγήσει κανείς με το αυτοκίνητο από τη Μάλτα μέχρι τη Στοχόλμη χωρίς να τον σταματήσουν ούτε μία φορά. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό που επιτεύχθηκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα σύνορα, όπως ξέρετε κατά παρελθόν, προκάλεσαν πολλούς πολέμους, όπως τα σύνορα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Γερμανία. ή τα σύνορα ανάμεσα στην Κορίτσια και τη Νέα Κορίτσια. Αυτά δεν είναι αφηρημένα. Αυτά που σας λέω είναι πολύ συγκεκριμένα και αυτό είναι απλώς ένα παράδειγμα. Ε, δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν υπάρχουν εμπόδια. Ένα από τα εμπόδια αναφέρθηκε από τον ε, κύριο Αγκουλιάρ είναι η αύξηση του λαϊκισμού, του εθνικιστικού λαϊκισμού με την αρνητική έννοια της λέξης. Δηλαδή προκαλούνται εμπόδια στην ελεύθερη μετακίνηση των ανθρώπων. Πολλοί λοιπόν λένε ότι καταβάλλονται προσπάθειες ε, να αποδομηθούν αυτά που επιτεύχθηκαν με πάρα πολλές θυσίες. Για μένα το σύστημα Schengen είναι ακρογωνιαίος λίθος. Ε, πρέπει να είναι σαφές αυτό. Ε, κατόπιν τούτου πρέπει να επαγρυπνούμε και δεν πρέπει να εισάγουμε μόνοι μας εμπόδια σε αυτό που κατά την άποψή μου είναι κληρονομιά για την επόμενη γενιά. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τους τρεις βουλευτές για τις ερωτήσεις τους όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος πριν από τρία χρόνια βεβαίως με τη Λισαβόνα και τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων που θέτουν τον πολίτη στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Αυτό ακριβώ ήταν και ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός. Από τον Φεβρουάριο του 2010 ξεκινήσαμε να υλοποιούμε αυτό το βήμα. Είναι η πρόεδρος η κυρία Ρέντινγκ, η οποία λόγω προσωπικού κολλήματο δεν μπορούσε να είναι σήμερα μαζί μα, αλλά και η επιτροπή ε, Μάλστρομ είχαν την ευκαιρία να συνδιαλεγούν με την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ για την ενδιάμεση αξιολόγηση του προγραμματό τη Στοκόλμης πέρσι τον Δεκέμβριο. Επιτρέψτε μου να σα θυμίσω μερικά από τα επιτεύγματα στον τομέα τη δικαιοσύνη. Σημείωσε μεσημερική πρόοδο στον τομέα της αστικής ε, δικαιοσύνη πούμε, την εσωτερική αγορά, την κίνηση δικαιοσύνη για την ανάπτυξη, το οποίο σημαίνει συγκεκριμένα μέτρα για να επανέλθει η Ευρώπη στον δρόμο της ανάπτυξης. Για παράδειγμα, εξαλείψαμε την δικασία executor. Οι αποφάσεις, οι δικαστικές αποφάσεις σε μια χώρα αναγνωρίζονται αυτομάτως σε μια άλλη χώρα μέλος. Επίσης, για την αφαιρεγγιότητα, το γνωστό πακέτο ενημερώνει τους ε, σχετικούς κανόνες. Θέλουμε οι βιώσιμες επιχειρήσεις να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία για να περισσώσουμε και τις θέσεις εργασίας. Το μεταρρυθμιστικό πακέτο για την προστασία των δεδομένων. Μειώνουμε έτσι τον διοικητικό φόρτο για τις επιχειρήσεις και τα πρόσωπα παρέχοντα ταυτόχρονα προστασία. Επίση στον τομέα τη ποινική δικαιοσύνη. είμαστε ιδιαίτερω υπερήφανοι για την πρόοδο που σημειώσαμε στην, στον τομέα τη προστασία των θυμάτων. Έχουμε τη σχετική οδηγία καθώ και τον σχετικό κανονισμό με τα οποία βελτιώνουμε την προστασία των θυμάτων κατά τη διάρκεια μια ποινική δική. Επίση ενισχύσαμε και βελτιώσαμε τις δικονομικές διαδικασίες, τα θέματα των μεταφράσεων, έχουμε επίσης μια οδηγία για το δικαίωμα στην πληροφόρηση. Προστατεύουμε καλύτερα επίσης τα θύματα σε όλη την Ευρώπη. Όλα αυτά είναι συγκεκριμένα επιτεύγματα τα οποία αφορούν τον απλό πολίτη. Χάρη στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο που θέλω να ευχαριστήσω για τις κοινές τους προσπάθειες. Πολύ σύντομα η οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο, σε νομική υποστήριξη θα είναι και αυτή έτοιμη. Είναι ένα θέμα το οποίο νομικός αλλά και διαδικαστικός ισχύει αλλά εφαρμόζεται με διαφορετικό τρόπο σε κάθε χώρα. Στον ποινικό τομέα προτείναμε ελάχιστη διαδικασία και ελάχιστε κυρώσει για να προστατεύσουμε τα οικονομικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και του Euro κατά τη παραχάραξη. Ο στόχο είναι απλός Να αξιοποιήσουμε την ποινική νομοθεσία για να ενισχύσουμε την προστασία των κοινών μα αγαθών. Καλούμε το Κοινοβούλιο να συνεργαστεί μαζί μα επί αυτού που θεωρούμε προτεραιότητα. Τα δικαιώματα των πολιτών αποτελούν θεμελιώδε ε, αγαθό σε αυτή την διαδικασία. Στα πλαίσια αυτά, τα, στα τέλη Μαου, θα παρουσιάσουμε την αξιολόγηση τη πρόοδου όσον αφορά το χάρτη και την έκθεση δικαιωμάτων ανδρών και γυναικών. Επίση την πρόοδο στην υλοποίηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Πέραν όμω αυτών, και πέραν και πέραν του προγράμματος της Στοκχόλμης που αποτελεί μια στρατηγική και μόνο κατεύθυνση, κάναμε και άλλα πράγματα. Δεν περιοριστήκαμε μόνο στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το λεγόμενο πίνακα επιδόσεων για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη να είναι πιο αποτελεσματικά στην παροχή αποτελεσματική δικαιοσύνη θέτουμε έτσι συγκεκριμένου στόχους, αξιολογούμε την πρόοδο και συγκρίνουμε τους στόχους, την ποιότητα και την αντικειμενικότητα της δικαιοσύνης σε όλα τα κατημέλη. Ορισμένοι αποκαλούν αυτό το σύστημα, σύστημα κατάδειξης ε, αυτών που υστερούν. Όμως εμείς το αντίθετο θέλουμε να εγκομιάσουμε αυτούς που τα καταφέρουν καλύτερα. Είμαστε υπερήφανοι επίση για τα επιτεύγματά μα στον τομέα του ασύλου. Στην επόμενη ολομέλεια το Κοινοβούλιο θα υπερψηφίσει μια πράξη για έναν χώρο ελεύθερο και ανοιχτό που θα παρέχει προστασία στα θύματα και όπου τα κρατημέλη θα συνεργάζονται επιδεινύοντας αλληλεγγύη. Επίσης το σύστημα θεωρήσεων του Schengen και το Schengen Information System, το σύστημα πληροφοριών Schengen και αυτά προχώρησαν. Έχουμε τα σωστά εργαλεία πλέον στα χέρια μας που εξασφαλίζουν ελεύθερη κυκλοφορία πέραν των συνόρων και το οποίο απολαμβάνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες και θα συνεχίσουν να απολαμβάνουν στην Υπηρό μας. Έχουμε επίσης ένα χώρο ελευθερίας για τους εργαζόμενους και για καλύτερη διακυβέρνηση του χώρου Σέγγεν, με καλύτερη επιτήρηση των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στα δύο είμαστε πιθανώς κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Επίσης, η Frontex έχει νέα εντολή για πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις, παρέχοντας διαβεβαιώσεις και διασφαλίσεις για τα θεμελιώδη δικαιώματα και η Europol επίσης έχει μια νέα εντολή για την εποχή μετά την Λισαβόνα. Έχουμε επίσης μια στρατηγική για την εσωτερική ασφάλεια και έχουμε και τακτικές εκθέσει για την εφαρμογή τη συνομολογήσαμε συνθήκε με τις ΗΠΑ Πολιτείες για την τρομοκρατία και για το PNR με την Αυστραλία. Άλλε οδηγίες επίσης αφορούν την αποφυγή κακοποίηση των παιδιών στο διαδίκτυο και έχουμε και, έναν, και νέα νομοθεσία όσον αφορά τους, τις πρόδρομες ουσίες για τα εκρηκτικά και θεσπίσαμε και ένα μηχανισμό παρακολουθήσει της παραγωγής αυτών των υλών. Επίσης ε, κινητικότητα και μετανάστευση. Ξεκινήσαμε συζητήσεις με πολλές γειτονικέ τρίτες χώρες. Σημειώσαμε πρόοδο στην διευκόλυνση έκδοσης θεωρήσεων και στις συμφωνίες επανεισδοχής. Επίσης έχουμε προτάσεις ε, για την ανταλλαγή ερευνητών και φοιτητών, ενδοτερικών εκπαιδευομένων και αναπτύσσουμε και μια ατζέντα για την ένταξη υπηκών τρίτων χωρών, καθώς και για την επανένωση των οικογενειών. Υπάρχουν ακόμα πολλά πράγματα που πρέπει να κάνουμε βεβαίω. Για παράδειγμα, αυτή τη στιγμή εργαζόμαστε εντατικά πάνω σε μια πρόταση για το Γραφείο Ευρωπαίου Εισαγγελέα για την αντιμετώπιση του εγκλήματο κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά τη ε, διαφθοράς, ασφάλεια στο διαδίκτυο. Όλα αυτά παραμένουν πρώτες προτεραιότητές μας. Δικαιοσύνη και εσωτερικές υποθέσεις. Και εδώ Πρόκειται έναν ευαίσθητο τομέα που παλαιότερα ήταν εθνικά αποκλειστικά αρμοδιότητα. Και όμως προσαρμοζόμαστε στις νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες και το νέο νομοθετικό πλαίσιο που προέκυψε από τη Λισαβόνα. Υποβάλαμε πολλές νομοθετικές προτάσεις, αλλά να τονίσω για άλλη μια φορά την σημασία της αποτελεσματικής υλοποίησης της σχετικής νομοθεσίας που ήδη βεβαίως έχουμε εγκρίνει. Μια συγκεκριμένη ανάγκη που συνειδητοποίησαμε τους τελευταίους μήνες αφορά το κράτος δικαίου. Και κλείνω με αυτό το σχόλιο. Όπως είπε και ο πρόεδρος Μπαρόσο, τους τελευταίους μήνες και συγκεκριμένα αυτό το είπε ο πρώτος Μπαρόσο πέρσι τον Σεπτέμβριο, είπε λοιπόν ότι χρειαζόμαστε καλύτερα εργαλεία, πιο αποτελεσματικά εργαλεία. Δεν θέλουμε μόνο άσπρο ή μαύρο. Ούτε θέλουμε το άρθρο 7 που είναι τα πυρηνικά μα όπλα, ούτε απλή δύναμη τη πυθού. Θέλουμε και διαμέση λύσει. και ελπίζουμε ότι το Κοινοβούλιο θα μα υποστηρίξει, λέει ο Πρόεδρο Μπαρόσο, για να θεσπίσουμε ένα νέο μηχανισμό ο οποίο θα δώσει τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να λαμβάνει κάθε φορά την απαραίτητη αποτελεσματική δράση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Κύριε Μπόρτς, ακολουθούν οι ομιλητές εξ ονόματος των πολιτικών ομάδων με πρώτο τον κύριο ε, Τσβίφκα για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε. Όταν πριν από τρία χρόνια ε, θεσπίσαμε το πρόγραμμα της Στοχόλμης και σε λεπτομέρειες, γνωρίζαμε ότι ήταν πάρα πολύ φιλόδοξο. Ήταν πολλές οι πρωτοβουλίες που χρειαζόταν ε, για θέματα δικαιοσύνης, ε, εμπορικό δίκαιο και αστικό δίκαιο. Ήταν δύσκολο να εφαρμοστούν και πώς να συναντηθούν 27 νομοθεσίες για να λυθούν τα πιο επίγοντα προβλήματα. Επιλέξαμε μια προσέγγιση για τους πολίτες μας που κυκλοφορούν ελεύθερα και επιλέγουν πού να εγκατασταθούν και πού να εργαστούν. Ε, είναι πολύ σκληρή η δουλειά αυτή, δεν διαφωνώ και πάρα πολύ απαιτητική από τεχνικής πλευράς. Ωστόσο, Βρυξέλλες 1, Ρώμη 3, ε, δεν είδαμε μεγάλες ε, πρόοδους εκεί. Το είπαν και άλλοι ομιλητές. Ορισμένα βήματα έχουν γίνει με τη προστιθέμενη αξία για τους πολίτες μας και για τις εταιρείες που έχουν διασυνοριακή δράση. Συμμετείχα σε πολλές ε, συσκέψεις ε, και κατάλαβα ε, ότι παρά τις καλές προθέσεις ορισμένων εκκρεμούν οι νομοθεσίες χρόνια ολόκληρα. Με το πρόγραμμα της Στοχόλμης ε, ξεκινήσαν ε, ορισμένες νομοθετικές διαδικασίες που ελπίζω να ευδοκιμήσουν προς όφελος των πολιτών. Γιατί καμιά φορά οι πολίτες βρίσκονται σε ε, δινή θέση και σε περίεργες καταστάσεις. Ε, όσοι εργάζονται λοιπόν στον τομέα της δικαιοσύνης θα πρέπει να γνωρίζουν τους νέους κανονισμούς ε, περί διαζυγίων, ε, κληρονομικών ζητημάτων και άλλων νομικών υποθέσεων. Ως μέλος της Νομικής Επιτροπής επανειλημμένα έχω τονίσει εδώ στο Κοινοβούλιο ότι ε, όταν υπάρχει άγνοια νόμου δεν εφαρμόζεται ο νόμος. Χρειάζεται λοιπόν η εκπαίδευση και ε, των νομικών και των δικηγόρων και των δικαστών. Πολύ συχνά εστιάζουμε σε δράσεις πληροφόρησης και ενημέρωση στους πολίτες. Θα πρέπει όμως να είμαστε πιο ανοιχτοί στην επικοινωνία μας και να ε, προβάλλουμε τις υφιστάμενες λύσεις ε, στο κοινοτικό δίκαιο, στο ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχει γίνει πρόοδος, αλλά περιμένουμε περισσότερο ακόμα για την αμοιβαία αναγνώριση, ας πούμε, διαφόρων πιστοποιητικών ε, και εγγράφων των κρατών μελών. Ε, είπαμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα χώρο ασφάλεια, ελευθερία και δικαιοσύνη και μέχρι να ολοκληρωθεί αυτό δεν θα έχει τελειώσει το πρόγραμμα τη Στοκχόλμη θα παραμείνουμε σε επαφή. Βεβαίω θα πρέπει να αξιοποιήσουμε πάντα τι ευκαιρίε που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν γίνει πολλά, απομένουν ακόμα πολλά. Δεν μπορούμε να επαναπαυθούμε στι δάφνε μα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα ε, δημοσίευσε μια πρωτοβουλία για ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών της Ένωσης που δείχνει ποια είναι τα επόμενα βήματα. Για το λόγο αυτό, τελειώνω Πρόεδρε, για το λόγο αυτό λοιπόν πιστεύω ότι ε, ε, χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια. Ευχαριστώ για δύο μισή λεπτά ο κύριος Γκερέρο Σαλόμ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Η νομιμοποίηση και η νομιμότητα των πολιτικών συστημάτων και εγχειρημάτων εδράζεται στα αποτελέσματα που παρέχει για να βελτιώνει την καθημερινότητα ε, των πολιτών, τη ζωή τους, αλλά και τις αρχές και τις αξίες που ενστερνίζονται και οι πολίτες. Και έτσι ε, χαρακτηρίζεται η πολιτική ένωση. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν δίνει καλά αποτελέσματα ε, ως προς την ανάπτυξη, ως προς την απασχόληση, ως προς τις δημόσιες πολιτικές στους πολίτες της. Και τι συμβαίνει με τις αξίες τώρα, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με ένα πολιτικό εγχείρημα που βασίζεται στην ελευθερία, που βασίζεται στην αλληλεγγύη, που βασίζεται στο σεβασμό των δικαιωμάτων αυτών των πολιτών της. Και η θεμελιώδης αξία είναι το αίσθημα του ανήκειν, να θεωρεί ο πολίτης ότι είναι τμήμα ενός πολιτικού σχεδίου κοινού, αλλά και ενός εδαφικού κοινού σχεδίου. Σε τρία χρόνια λοιπόν μάλλον τρία χρόνια μετά από το πρόγραμμα της Στοκχόλμης έγιναν πρόοδοι και αναφέρθηκε σε αυτό και ο Επίτροπος και ο Υπουργός. Αλλά θα ήθελα να τονίσω τρεις τομείς όπου υπάρχουν ακόμα προβλήματα. Πρώτον, η ελεύθερη κυκλοφορία. Ο Επίτροπος μας είπε ότι μπορεί από τη Μάλτα να φύγει αυτοκίνητο και να πάει στη Στοχόλμη χωρίς κανένα φραγμό, κανένα έλεγχο στην ελευθερία κινήσεων. Ναι, αυτό όμως γιατί γίνεται. Φαίνεται δεν έχετε πάει στη Δανία πρόσφατα από τη Γερμανία γιατί θα σας είχαν σταματήσει ή από την Ανατολική Ευρώπη κάποιο που θέλει να πάει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Γιατί και εκεί θα σα είχαν σταματήσει και εκεί μπαίνει τροχοπέδι στην ελευθερία κινήσεων. Γνωρίζουμε ότι στο Σέγγεν υπάρχει σύγκρουση για το θέμα αυτό μεταξύ Κοινοβουλίου και Συμβουλίου και επίση ξέρουμε ότι είναι πολύ δυσίωνε οι προβλέψει για την κυκλοφορία την ελεύθερη του Σέγγεν. Δεύτερο τομέα, η διαφάνεια. Παραμένει άλυτο το θέμα τη πρόσβαση στα έγγραφα. Και εδώ σε τούτη την Ολομέλεια κατατέθηκε προφορική ερώτηση για την εμπλοκή ε, στην οποία έχουμε ε, πέλθει. Προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών. Το τρίτο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο της Ευρώπης για τη Σύμβαση και καλό το Συμβούλιο και τους παροτρύνω αυτή στιγμή αποφανθεί το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων να ολοκληρώσουμε αυτή τη διαδικασία και να προστατεύσουμε καλύτερα τα δικαιώματα των πολιτών μας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γκερέρο Σαλόμ και τώρα για δύο λεπτά η κυρία Βίξτρομ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντικό το ότι μπορούμε να συζητήσουμε σήμερα το απόγευμα το θέμα αυτό μαζί σας το πρόγραμμα της Ευρώπης σε προάγει μια ανοιχτή Ευρώπη με τον πολίτη στο επίκεντρό της. Ε, πρέπει να αναλύσουμε το τι ακριβώς έχει γίνει και το τι πολύπεται ακόμα στο πρόγραμμα μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι πρέπει να υπάρχει ένα κοινό σύστημα χορήγησης ασύλου. Έχουμε επιτύχει λοιπόν ε, κυρίως σε μια εποχή όπου οι οικονομίες ε, των κρατών μελών χυμάζονται κατορθώσαμε να επιτύχουμε σημαντική πρόοδο και πρέπει να σας πω ότι είμαι ιδιαίτερα ευτυχής για το ότι έχουμε πλέον νομική ασφάλεια για τους ετούντες άσυλο. Αυτό λοιπόν προσδίδει στην αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη και θα βελτιωθεί η κατάσταση περαιτέρω στο μέλλον. Στο πρόγραμμα προβλέπεται η εντατικοποίηση του προγράμματος ε, ε, εγκατάστασης των προσφύγων ε, και κυρίως και των προσφύγων του οποίους προστατεύει η αρμοστία των Ηνωμένων Εθνών. Αναφερθήκατε στην μετανάστευση εργαζομένων. Εγώ ήμουνα εισηγήτρια ε, για, τις, ε, για θέματα ερευνητών που έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό λοιπόν το θέμα πρέπει πλέον να αντιμετωπιστεί. Οφείλουμε να σταματήσουμε τον, την ε, αφέμαξη επιστημονικού δυναμικού και θέλω να τελειώσω υπενθυμίζοντας στον Επίτροπο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υποσχεθεί να καταθέσει μία πρόταση για την αμοιβαία αναγνώριση τις θέσεις του πολίτη. Ακόμα δεν έχει γίνει κάτι συγκεκριμένο. Ε, διακόπηκε η ομιλήτρια, η κυρία Σαρτζεντίνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ακούω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο ε, να παριθμούν ένα κατάλογο προγραμμάτων στο Στοκχόλμη, στο χώρο ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης και μάλιστα τα πεπραγμένα αυτά δηλώνεται ότι είναι επιτυχή. Εντάξει, αλλά δεν μετράμε ε, μόνο την κατάσταση στην Ένωση, ε, στην οικονομική κρίση και στις χρηματαγορές, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο γίνονται διάφορες συζητήσεις στην Ένωση για την ηθική, τη δεοντολογία, τα δικαιώματα των πολιτών, τα δικαιώματα των υπόπτων, τα δικαιώματα των ε, προσφύγων και πώς γίνεται η συζήτηση στο Συμβούλιο. Το Κοινοβούλιο εδώ και χρόνια είναι έτοιμο και περιμένει αυτό που προσεχώς θα ψηφίσετε για το άσυλο και τη μετανάσκευση. Και το Συμβούλιο σπαράζεται από ε, διάφορες ε, μάχες και δεν μπορούν να βρουν τα κράτη μια λύση. Ήταν πριν τη συνθήκη της Λισαβόνας το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Νομίζω δεν θα πρέπει να κάνουμε τόσο μεγάλα προγράμματα στο μέλλον. Ε, θα πρέπει να έχουμε ισόρροπη νομοθεσία ε, με ε, το βλέμμα στραμμένο στα θεμελιώδη δικαιώματα, όχι μόνο στο ποινικό δίκαιο, αλλά και η διακυβερνητική συνεργασία να μην είναι ένα ενιαίο ε, πρόγραμμα που να τα περιλαμβάνει όλα, ψηφίδα-ψηφίδα. Σιγά-σιγά έχουν ξεπεραστεί αυτά τα συστήματα. Επίσης δεν μπορούμε να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο στο βαθμό που το Συμβούλιο δεν μπορεί να συμφωνήσει. Και πραγματικά είναι κραυγαλαίο το παράδειγμα της αμοιβαία εμπιστοσύνη στην ποινική συνεργασία. Ε, ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης είναι κάτι ε, που ε, μεταφέρει πολίτες από τη μια χώρα στην άλλη οι οποίοι μετάγονται χωρίς να έχουν την κατάλληλη προστασία και χωρίς να γνωρίζουν τα δικαιώματά τους. Αυτό που κυριαρχεί τώρα είναι η αμοιβαία κάχη υποψία και δυσπιστία. Ποιο είναι το μέλλον της Ευρώπης έτσι. Θα πρέπει να εμπιστευόμαστε ένας τον. Εντάξει, σταματώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Σαρχεντίνη. Και τώρα για δύο μισή λεπτά ο κύριος Κίρκοπ. Πρόεδρε, βρισκόμαστε ε, στο τέλος αυτής της θητείας όπου το Κοινοβούλιο έχει πλέον νέες αρμοδιότητες υπήρξαν επιτυχίες και αποτυχίες η δική μου άποψη δεν έχει αλλάξει εγώ εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε λιγότερα αλλά καλύτερα ε, και αυτό αφορά την ε, ε, το κυβερνό έγκλημα, όπως επίσης ε, και τους ασυνόδευτους ανήλικους ε, που είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη. <clears throat> Πρέπει να είμαστε φιλόδοξοι αλλά και ρεαλιστέ γιατί μπορούμε να πετύχουμε. Καλό το Κοινοβούλιο και την Κομισιόν να στοχεύσουν εκεί που μπορούν να πετύχουν τα περισσότερα με σαφήνεια αντί για περίπλοκες καταστάσεις. Εάν λοιπόν υπάρχει καλύτερη εμπιστοσύνη και συνεργασία και αποτελεσματικότητα, αν η Κομισιόν μπορεί να διασφαλίσει όλα αυτά, τότε θα υπάρχει ένα σύστημα όπου στα κράτη-μέλη ναι, θα υπάρχουν διαφορετικά νομικά συστήματα, αλλά αποτελεσματά ουσιαστικά. Ε, το θέμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας ε, δεν νομίζω ότι είναι η μόνη λύση. Ε, δεν έχουν υπάρξει καμία αναθεώρηση τα τελευταία χρόνια και μπορούμε να πετύχουμε καλύτερα αποτελέσματα μέσα από τη συνεργασία ανάμεσα στους ε, θεσμούς. Η ε, αναθεώρηση όμως που είναι απαραίτητη δεν έχει λάβει χώρα. Καλό λοιπόν την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αξιολογήσει τις επιτυχίες και τις αποτυχίες του προγράμματος της Στοχόλμης για να προχωρήσουμε επικοδομητικά αλλά όχι στα τυφλά. Ευχαριστώ πολύ. Ε, επιτρέπει μια ερώτηση από τον συνάδελφο Ντάρτμοθ. Oh, ναι. Βεβαίως, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο. Κύριε Κέρκοπ, εσείς πιστεύετε ότι το Ρωμένο Βασίλειο θα πρέπει ε, να ε, ζητήσει opt-out του χρόνου που θα έχει την ευκαιρία από το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ναι ή όχι. Να εξαιρεθεί. Σας ευχαριστώ ε, αξιότιμε συνάδελφοι για την ερώτηση. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα αξιολογήσει τη θέση για όλα τα θέματα και μεταξύ αυτών και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, τα υπέρ και τα κατά του και την ανάγκη μεταρρύθμισης του. Υπάρχουν πολλοί άλλοι εδώ που θα συμφωνήσουν μαζί μας ότι χρειάζεται μεταρρύθμιση, αλλά χωρίς να υπολογίζει κανείς ε, την πλήρη επίδραση και τις επιπτώσεις σε όλους και τους πολίτες της ε, ε, Ηνωμένου Βασιλείου αλλά και τους υπολείπους, δεν μπορούμε από τώρα να σας πούμε τι θα κάνουμε, να περιεξοφλήσουμε το μέλλον για αυτό το θέμα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Κέρκοπ. Και τώρα για 1,5 λεπτό ο κύριος Τριανταφυλλίδης παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, για την προετοιμασία του επόμενου πολιετούς προγράμματος για το χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης δεν αρκεί μια απαρίθμηση των προτάσεων που υπέβαλε η Επιτροπή ή που εγκρίθηκαν από τους συνομοθέτες, αλλά απαιτείται ένας γνήσιος ποιοτικός και όχι μόνο ποσοτικός έλεγχος είναι αναγκαίο να αξιολογήσουμε το πού βρισκόμαστε σε σχέση με το δίλημα δικαιώματα ή ασφάλεια. δική μας εκτίμηση είναι ότι σημειώνεται πάντοτε πρόοδος στα θέματα ασφάλειας όπως για παράδειγμα στο swift ή τα smart borders αλλά η διαδικασία αργεί αισθητά όταν πρόκειται για θεμελιώδη δικαιώματα όπως το access to documents ή το data protection. μια τέτοια τάση έχει τη σημασία της καθώς οι προτάσεις που σχετίζονται με την ασφάλεια είναι πάντα εξωφρενικά ακριβές. θα μπορούσατε αλήθεια κύριε επίτροπε να μας πείτε ποιες πολιτικές θα πρέπει να υποβαθμιστούν περαιτέρω στο επόμενο πρόγραμμα για να καταστεί δυνατή η χρηματοδότηση της πρότασης για τα smart borders. αυτός ο ποιοτικός έλεγχος πρέπει επίσης να αξιολογήσει τις νέες διαθεσμικές διευθετήσεις που εισήγαγε η συνθήκη της λισαβόνας όσον αφορά τη δημοκρατική νομιμότητα με βάση την εμπειρία μας το κοινοβούλιο παραμελείται συστηματικά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων προκειμένου να διασκεδαστούν οι ανησυχίες των κρατών μελών στο συμβούλιο. χρειάζεται να υπενθυμίσω ότι προκειμένου να ξεπεραστεί το αδιέξοδο στο συμβούλιο σχετικά με το eurodac η επιτροπή παρουσίασε νέα πρόταση αγνοώντας πλήρως τη θέση πρώτης ανάγνωσης του κοινοβουλίου. Ευχαριστώ πολύ κύριε Τρεταφυλλίδη. Και τώρα για ένα λεπτό το λόγο έχει ο συνάδελφος Ζέλστρα. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Πρόεδρε, ερωτώ, τι το καλό έχει το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Το πρόγραμμα είναι κατά των συνοριακών ελέγχων που θέλουν να κάνουν οι χώρες για να αφήσουν τους εγκληματίες εκτός. Το πρόγραμμα δέχεται ε, το να είναι αδύνατο ε, κανείς να αντιταχθεί στο ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και ε, ε, άδικα φυλακίζονται πολλοί πολίτες της Ένωσης σε κελιά του εξωτερικού ποινικό δίκαιο. Πού είναι η εθνική κυριαρχία των κρατών μελών. Η κοινή πολιτική ασύλου δεν οδήγησε σε μείωση της εξάπλωσης των μεταναστών, απλώς ε, συσσόρευση και συγκέντρωσή τους σε κάποια κράτη-μέλη. Συμπέρασμα, το πρόγραμμα δεν είναι ε, προς όφελος των πολιτών, το αντίθετο. Το κομβικό ζήτημα θα πρέπει να είναι εάν εξυπηρετείται ο πολίτης από το πρόγραμμα της Σοχόνης. η δική μου απάντηση είναι αρνητική. Ε, είναι αποτυχία αυτό το πρόγραμμα να ε, εκπνεύσει και να μην αντικατασταθεί από άλλο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ζέλστρα και τώρα για τρία λεπτά ο κύριος Παπα-Νικολάου παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Στο ερώτημα χρειαζόμαστε ένα νέο πρόγραμμα σε αυτή τη φάση μετά το πρόγραμμα της Στοχόλμης νομίζω η απάντηση είναι καθαρή. Το πρόγραμμα της Στοχόλμης ήταν και παραμένει φιλόδοξο ήταν και παραμένει σημαντικό να εφαρμοστεί. Και στο σημείο αυτό θέλω να συμφωνήσω με αυτά που υπόθηκαν και από το Συμβούλιο και από την Επιτροπή και βεβαίως να τονίσω ειδικά σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση της αξιότιμης κυρίας Υπουργού ότι δεν αρκεί να λέμε ότι οι Υπουργοί έδειξαν ικανοποίηση και προσδοκούν περισσότερα συνέχεια. Έχει πολύ μεγάλη σημασία και η κριτική για όσα δεν έγιναν, για όσα καθυστέρησαν, η κριτική για την εφαρμογή των πεπραγμένων και των αποφάσεων που λαμβάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο δεν υπάρχει αμφιβολία ότι σημαντικά νομοθετήματα έχουν προχωρήσει έχουν ολοκληρωθεί δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι η κατάσταση σήμερα η διαθεσμική λειτουργία σε σχέση με αυτή που είχαμε το 2008 ήταν είναι σήμερα κατά πολύ αναβαθμισμένη η συνθήκη της Λισαβόνας αλλάζει το πλαίσιο λειτουργίας όλων μας σε αυτό προσαρμοζόμαστε ακόμα τα τρία χρόνια αυτά είχαμε πολύ σημαντικές εξελίξεις. η συνήθι νομοθετική διαδικασία πλέον που είναι η συναπόφαση νομίζω ότι λειτουργεί ολοένα και καλύτερα. βεβαίως όμως έχουμε και σημαντικές ελλείψεις και σημαντικά κενά τα οποία πρέπει να εκπληρώσουμε. δεν είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα έχουμε καταλάβει ότι έχουμε απόλυτη ανάγκη να έχουμε συμφωνία για το επόμενο διάστημα στις κοινέ προκλήσεις που χρειαζόμαστε σε ευρωπαϊκό επίπεδο και σε αυτό να συμφωνεί και η επιτροπή και το συμβούλιο και βεβαίως και το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο. η ισορροπημένη προσέγγιση σε όλα τα θέματα είναι καθοριστική. χρειαζόμαστε στα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε τώρα την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη ασφαλώς και το δικαίωμά του στον ιδιωτικό του χώρο χρειαζόμαστε όμως και ασφάλεια χρειαζόμαστε τα δικαιώματα στο πακέτο ασύλου των μεταναστών και των ετούντων άσυλο χρειαζόμαστε όμως και καταπολέμηση της παράνομης μετανάστευσης. κυρίες και κύριοι συνάδελφοι την περίοδο αυτή καταγράφεται από τις ευρωπαϊκές μετρήσεις ότι οι ευρωπαίοι πολίτες νιώθουν λιγότερο ασφαλείς από ό,τι στο παρελθόν και σε αυτό ακριβώς το αίσθημα των ευρωπαίων πολιτών έρχεται η άνοδος του εξτρεμισμού σε πολλά κράτη μέλη αναφέρθηκε ήδη ακόμα και σε εκείνα που δεν πλήττονται το ίδιο σφοδρά από την κρίση και αυτό είναι μια ακόμη μεγάλη πρόκληση για την ασφάλεια και την ελευθερία. θα πρέπει και αυτό να το δούμε. αναφέρθηκε η κυρία υπουργό στη ρήτρα της αλληλεγγύης. την αναφέρουμε συνέχεια τη ρήτρα και χθε είχαμε μια σχετική συζήτηση για το πρόγραμμα εσωτερικής επανεγκατάστασης. σε πολλά ζητήματα όμω, η ρήτρα αυτή παραμένει απλώ θεωρία και δεν έχουμε προχωρήσει στην πράξη. Κυρίες και κύριοι, φέτος το 2013 έχει χαρακτηριστεί ως ευρωπαϊκό έτος για τους πολίτες της Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι στο χέρι μας και στο χώρο της ασφάλειας, ελευθερίας και δικαιοσύνης να έχουμε στο κέντρο μας σε ό,τι κάνουμε τον πολίτη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παπα-Νικολάου. Και τώρα για μισή λεπτά το λόγο έχει η κυρία Γκυγιόμ. Το πρόγραμμα του Τάμπερ το 1999 και της Χάγης το 2004 έτσι, και το πρόγραμμα της Στοκχόλμης είναι φιλόδοξο. Αλλά μας αφήνει μια πικρία η ενδιάμεση αναθεώρηση. Ε, πτέθηκε σε ε, ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνης και τόσα χρόνια μετά είναι σαν να είμαστε στη συνθήκη του Μαστρίχτ όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήταν απλώς συμβουλευτικό όργανο ε, και απότερο ε, το βλέμμα των άλλων θεσμικών οργάνων προς το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να καταλάβουν τα θεσμικά όργανα και το Συμβούλιο ιδιαίτερα ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα. Και λέω ότι είναι μια πικρία γιατί εξαρτώμαστε από την στρατηγική για την ιστορική ασφάλεια, τη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων. Αυτά είναι σημαντικά θέματα για τους πολίτες και έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς ή σε άλλα δίκτυα που στερούνται δημοκρατικού ελέγχου. Επίσης, η αλληλεγγύη, η αλληλεγγυη διακρατική είναι στο άρθρο 80 της συνθήκης αλλά παραμένει νεκρό γράμμα. Ε, Πού είναι το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου, το κοινό. Δυσκολευόμαστε πάρα πολύ και δείχνει ότι η διακυβερνητική προσέγγιση κυριαρχεί ακόμα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ε, ο απολογισμό λοιπόν και τα αποτελέσματα είναι μάλλον ανεπαρκή. Έχουμε συγκεκριμένους στόχου και σημαντικούς όπως είναι η οδηγία κατά των διακρίσεων, καμία πρόοδος, είναι κατάφορο παράδειγμα αυτό. Και αγαπητοί συνάδελφοι και κύριε Επίτροπε, θέλαμε να μας μιλήσετε και για την ενίσχυση ε, της αξιοπιστίας αυτών των ευρωπαϊκών οργάνων και τι προσπάθειες καταβάλλετε προς την κατεύθυνση αυτή. Ευχαριστούμε πολύ. Για ένα λεπτό, ο κύριος ε, Βοσικόψκι. Κύριε Πρόεδρε, Εγώ επειδή το κόμμα μου αποκαλείται νόμος και δικαιοσύνη χαίρομαι πάρα πολύ που μία από τις προτεραιότητες του προγράμματος Στοκχόλμης, Στοκχόλμης είναι ακριβώς ο νόμος και η δικαιοσύνη. Στην Ευρώπη μου φαίνεται έχουμε επάρκεια νόμων και ε, έλλειψη δικαιοσύνης. Βεβαίως η δικαιοσύνη δεν είναι αλάθητη και το λέω αυτό με βάση τις εμπειρίες από τη δική μου τη χώρα αλλά και γνωρίζοντας και το τι συνέβη σε άλλες χώρες. Μιλάω για περιπτώσεις περιπτώσεις όπου είχαμε απαγωγή παιδιών, απομακρύνθηκαν τα παιδιά από τους γονείς τους. Η δικαιοσύνη πρέπει να είναι ανεξάρτητη, αλλά ε, δεν μπορεί να είναι και υπεράνω του δημοκρατικού ελέγχου. Η δικαιοσύνη δεν μπορεί να γίνει κράτος εν κράτη και αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πολύ περισσότερο. Ευχαριστούμε για ένα λεπτό, η κυρία Έρνστ. Ευχαριστώ πολύ. Ε, θα ήθελα να πω το εξής. Ε, ε, είναι πραγματικά εντυπωσιακό το τι ακούμε σήμερα εδώ, κυρίως όταν πρόκειται για την αξιολόγηση του δικού τους του προγράμματος. Και πραγματικά δεν υπήρξε καμία ουσιαστική αξιολόγηση. Ο πιο απλός ε, υπουργός ε, στα δικά μας ε, τα κράτη-μέλη θα προσπαθούσε περισσότερο, κυρίως διότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση βλέπουμε ότι πολλοί επιτρέπουν πράγματα που είναι ανύπαρκτα. Όταν προκύπτουν όλα αυτά τα δαπανηρά εργαλεία χωρίς ποτέ να έχει γίνει αξιολόγηση των παλαιότερων κατά πόσον ε, έχουν εκπληρώσει τους στόχους τους. Ε, αυτό μοιάζει ότι δεν ενοχλεί κανένα, δεν ενοχλεί ούτε την Κομισιόν ούτε το Συμβούλιο όταν το Smart Border ε, Register πρόγραμμα ε, που είναι πολύ δαπανηρό ε, τελικά δεν υλοποίησε το στόχο του. Διακόπηκε η ομιλήτρια για 1,5 λεπτό. Ο συνάλφος κύριος Εγενχάουζε έχει το λόγο. Κρίμα που διακόψατε την κυρία Έρνστ. Νομίζω αυτά που είπε ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να πω το εξή, ότι όσον αφορά τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και πληροφοριών ε, για τα σωστά άτομα, τη συγκεκριμένη στιγμή, ε, την προστασία των δεδομένων, το δικαίωμα στην ιδιωτική σφαίρα. Όλα αυτά είναι κάποια κριτήρια για να δούμε αν επιτυχαίνει ε, το πρόγραμμα της Στοχόλμης ε, και συγκεκριμένα όσον αφορά τη διαχείριση των πληροφοριών. Η συνέπεια λοιπόν είναι σημαντικός στόχος του προγράμματος της Στοχόλμης. Υπάρχουν κάποιες πρωτοβουλίες, πλατφόρμες όπου ανταλλάσσονται οι πληροφορίε αναλύονται. Έχουμε επίσης τη στρατηγική για την διαχείριση της πληροφορία και αυτή ακριβώς είναι η ερώτησή μου προς το Συμβούλιο και προς την Επιτροπή. Δηλαδή το ερώτημά μου είναι αυτή η στρατηγική για τη διαχείριση της πληροφορίας έχει εφαρμοστεί στην πράξη και αν ναι, τι έχουμε επιτύχει. Θα ήμουν ευγνώμων αν μπορούσατε να μας ενημερώσετε λιγάκι από αυτού. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ τον συνάλφο κύριο Χάουζερ, Η κυρία Έρνστ ε, φαντάζομαι θα ευχαριστήσει για τα λουλούδια που πήρε από την άλλη πλευρά. Κοιτάξτε, ε, δική μου δουλειά δεν είναι ένα αξιόλογο ε, αν είναι καλές ή ε, όχι οι παρεμβάσεις, παρά μόνο αν τηρείται ο χρόνος αγόρευσης. Η κυρία Αντζελίλη για δύο λεπτά. Το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης ε, είναι μια πολύ σημαντική στρατηγική με συγκεκριμένες πράξεις ε, για να εφαρμοστεί στο συγκεκριμένο ευρωπαϊκό χώρο. Έχει σχέση με την ελευθερία, την ασφάλεια, τη δικαιοσύνη, όλα αυτά στην υπηρεσία του πολίτη. Καθορίστηκε ως πρόγραμμα δράσης το 2010. Ήταν ένα πρόγραμμα ιδιαίτερα φιλόδοξο. Ο στόχος ήταν να ε, προσφερθεί η μέγιστη δυνατή προστασία στις αξίες όπως σεβασμός για τον άνθρωπο, ανθρώπινη αξιοπρέπεια, ισότητα, αλληλεγγύη και παράλληλα στο κέντρο να μπει ο πολίτης ε, η καθημερινότητά του. Μπορούμε λοιπόν, κατά την απόψή μου, να κάνουμε ένα θετικό πρώτο απολογισμό. Αναφέρουμε παραδείγματος χάρη στην οδηγία ε, για την προστασία της τάξης στην Ευρώπη. Αυτό είναι ένα πρωτοπόρο εργαλείο. Αναφέρομαι στην οδηγία για τα δικαιώματα ε, των θυμάτων εγκλημάτων και αναφέρομαι επίσης ε, και στα διάφορα μέτρα που ελήφθησαν για την προστασία των ανηλίκων συμπεριλαμβανομένης και της οδηγίες περί ε, κακοποίησης και ε, πορνογραφίας ε, online. Εκεί ήμουν μάλιστα και η εισηγήτρια. Υπολείπονται βέβαια ακόμα πάρα πολλά και γι' αυτό θα ήταν χρήσιμο να υπάρξει μια αξιολόγηση ακριβώς για να μπορέσουμε να μετρήσουμε όλες τις δυσκολίες που έχουν προκύψει κατά την εφαρμογή. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσουμε να προβούμε στι απαραίτητες διορθώσεις, να ξεκινήσει μια νέα φάση, μια βελτιωμένη ε, συνεργασία για να χαρακτεί η σωστή στρατηγική από πλευράς κρατών μελών. Ευχαριστώ για 1,5 λεπτό η κυρία Γκέμψ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, η συνθήκη της Λισαβόνας έχει επιφέρει μείζονες αλλαγές ε, στη διαδικασία λήψης αποφάσεων σε αυτούς τους τομείς. Δεν βλέπουμε όμως την πράξη τα αποτελέσματα, ούτε την προσήλωση ε, των κρατών μελών να εκτελούν όλα αυτά που αποφασίζονται. Με βασικότερα παραδείγματα τη διακυβερνητική συνεργασία. Εκεί λαμβάνονται αποφάσεις. Οι Ρωμά αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα, δεν αναγνωρίζονται τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα παντού, ε, ούτε τα πιστοποιητικά τους και μια ε, κοινότητα κρίσιμη και ένας πληθυσμός στον οποίο θα μετρηθεί η δυνατότητα δημιουργίας χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Χρειάζεται αμεσότερη δράση στον τομέα αυτό και να διασφαλιστούν και τα θεμελιώδη δικαιώματα και αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε πολύ μεγαλύτερη αφοσίωση και προσήλωση από τα κράτη-μέλη στην υπόθεση αυτή. Και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζητούμε να δώσει ε, μια απάντηση στεναρή και πληρωμένη σε οποιοδήποτε αποπειράται να καταλύσει τις θεμελιώδεις αρχές και αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκιόνης και τώρα για ένα λεπτό η κυρία Βερζιά. Πρόεδρε, μπορούμε να προβούμε σε μια αξιολόγηση του προγράμματο μεταξύ των Ευρωπαίων που ψήφισαν το Μάστριχτ που πίστεψαν στην πρόοδο που υποτίθεται ότι αποτελούσε για την κοινωνική δικαιοσύνη. Είδα την πρόοδο που σημειώσαμε στη δεκαετία του 90, είδα το πρόγραμμα του Τάμπερεν, όμως από το 2000 και μετά είναι μάρτυρες μιας συλλογής πορείας. Η ασφάλεια υπερκέρεσε τα δικαιώματα. Με τη Λισαβόνα κάποιοι πίστεψαν ότι με την εσωμάτωση του χάρτη τα πράγματα θα άλλαζαν. Ελπίσαμε, όντως. Και πού βρισκόμαστε σήμερα. Οι περισσότερες πρωτοβουλίες σταματούν στο Συμβούλιο. Το δικαίωμα στο άσυλο, είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα και δείτε τι γίνεται με τους πρόσφυγες, με τους ε, πρόσφυγες, με τους μετανάστες στα σύνορά μας. Τα θεμελιώδη δικαιώματα, η δικαιοσύνη γνωρίζουν χειρότερες μέρες στην Ευρώπη, ιδιαίτερα για τους πλέον ευπαθείς. Ας αλλάξουμε λοιπόν κατεύθυνση, αν θέλουμε οι Ευρωπαίοι πολίτες να πιστέψουν και πάλι στο ευρωπαϊκό όνειρο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βαζιά και τώρα για δύο λεπτά κύριε Ματσόνη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Αυτή τη συγκεκριμένη περίοδο η Ευρωπαϊκή Ένωση παραπέει ε, στις ε, αναταραχές της οικονομικής κρίσης. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε μία απάντηση στους ε, πολίτες οι οποίοι νιώθουν ανασφαλείς και να τοποθετηθούμε πάνω στη διαδικασία της ολοκλήρωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να απαντήσει στις επιθέσεις της αγοράς και η απάντηση είναι η μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Η ε, πολιτική ένωση βέβαια δεν μπορεί να επιτευχθεί αν δεν υπάρχουν ε, εχέγγυα προς τον Ευρωπαίο πολίτη για το ότι έχει τα ίδια δικαιώματα και τις ίδιες υποχρεώσεις. Αν δεν εγγυηθούμε σε όλους τους πολίτες ένα δίκαιο σύστημα προστασίες προστασίας και παράλληλα αν δεν του προσφέρουμε τα μέσα ε, για να έχει την σωστή ε, δικαστική και νομική προστασία. Γνωρίζω πολύ καλά πόσο εργάστηκε η Επιτροπή, μπόρεσα να το παρακολουθήσω, ε, παρακολουθώντας τη δουλειά της κυρίας Ρέντινγκ και σήμερα άκουσα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση την παρέμβαση του Επιτρόπου Μπόρκ. Είμαι λοιπόν πεπισμένη ότι όλα αυτά τα οποία άκουσα έχουν τεθεί επιτάπητος. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχουν ακόμα υλοποιηθεί πάρα πολλά. Είμαι πρόεδρος Επιτροπής Αναφορών και ζω καθημερινά τη σχέση με τους πολίτες. Μπορώ λοιπόν να σας πω ότι ζω το πλεονέκτημα ε, αυτής της ειδική θέσης, της πλεονεκτικής θέσης, γιατί μέσα από το δικό μας το παρατηρητήριο παρακολουθούμε τι ακριβώς γίνεται και μπορώ να σας πω ότι είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το να υπάρχει ένας κοινός ευρωπαϊκός χώρος ελευθερίας, ε, δικαιοσύνης, ισότητα αναφέρω κάποια συγκεκριμένα παραδείγματα. Σε επίπεδο δικαιωμάτων έχουμε ζευγάρια ε, από διαφορετικές χώρες που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν ε, προβλήματα λόγω του ότι υπάρχουν εθνικιστικές απόψεις. Υπάρχουν ε, επίψεις περιπτώσεις ανθρώπων που δεν μπορούν να ξεπεράσουν τους φραγμούς. Πολλές φορές οι πτυχιούχοι δεν βρίσκονται στην ίδια φάση, στο ίδιο επίπεδο. Οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να μεταφέρουν τα εργασιακά τους δικαιώματα, τα στεξιωτικά τους δικαιώματα σε ένα άλλο κράτος. Υπάρχει λοιπόν έλλειψη προστασίας, διακόπτεται η ομιλήτρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Ρέγνερ για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμη κυρία Υπουργέ, αξιότιμη κυρία Επίτροπε. Το πρόγραμμα δράσης για την υλοποίηση του προγράμματος Σχόλμη έχει έρθει σε μια φάση πλέον αποφασιστική. Το είπατε κι εσείς κύριε Πίτρο, ολοκληρώθηκε η φάση Βρυξέλλε 1. Η προστασία ε, των δεδομένων ε, είναι ένα θέμα πάρα πολύ φλέγων. Η προστασία ε, και η αναγνώριση των πιστοποιητικών και των εγγράφων το ίδιο. Θα μας παρουσιάσετε λοιπόν μια έκθεση, ένα αποδεικτικό επιτυχίας. Αυτό που με ενδιαφέρει ιδιαίτερα είναι η οδηγία κατά των διακρίσεων. Στο πρόγραμμα της Στοχόλμης πραγματικά έχουμε ως πυρήνα του προγράμματος ε, προβλέψει ότι η ξενοφοβία, ο ρατσισμός, η ομοφιλοφιλοφοβία θα πρέπει να καταπολεμούνται. Δεν υπάρχουν όμως αντίστοιχες νομοθετικές προτάσεις. Τι γίνεται στο Συμβούλιο όμως και στην Επιτροπή όταν πρόκειται για την οδηγία κατά των διακρίσεων. Ένα άλλο θέμα, πολύ σημαντικό, το ανέφερε ο συνάδελφος Μπερλιγκουέ, η εφαρμογή, η υλοποίηση των συγκεκριμένων μέτρων. Οι πολίτες, άντρες και γυναίκες, συχνά αγνοούν ε, τα όσα έχουμε επιτύχει. Υπάρχουν ε, ε, πρωτοβουλίες για την ποινική δικονομία για την προστασία των πολιτών. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό και εμένα με ενδιαφέρει να μάθω πώς θα βελτιώσει την ενημέρωση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και ένα τελευταίο ερώτημα αφορά το διάλογο με την κοινωνία των πολιτών. Τι προβλέπετε με αλφαγιώτα εδώ και με ποιο τρόπο ε, επιλέγονται οι συνομιλητές μας εκπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών. Ευχαριστώ κυρία Ρέγνερ. Για δύο λεπτά ο κύριος Δίας Δεμέρα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχει αναθεωρηθεί ε, το πρόγραμμα ε, της Στοκχόλμης. Εγώ θέλω να αναφερθώ σε τρεις στόχους που δεν έχουν ακόμα επιτευχθεί και έχουν να κάνουν με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και της βαριάς εγκληματικότητας. Πρώτον, δεν έχει αναπτυχθεί το άρθρο 75 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς ε, το πάγωμα των στοιχείων ενεργητικού και τη χρήση ε, καταλόγων τρομοκρατικών οργανώσεων εσωτερικών στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτό δεν έχει αναθεωρηθεί από το 2009. Δεύτερον, απουσία νομοθετικών πρωτοβολιών σχετικά με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας. Τρίτον, και αυτό είναι πραγματικά πρόσφατο γεγονός και πάρα πολύ λυπηρό. Ε, το Ευρωπαϊκό PNR διακόπησε πρώτη ανάγνωση. Εγώ είμαι απεσιόδοξος ως προς τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Αλλά το πιο σοβαρό, κύριε Πρόεδρε, αφορά την έλλειψη ε, διοργανικής συμφωνίας. Σε τι αναφέρομαι και τι εννοώ. Εννοώ τη χρήση Μάλλον να το πω αλλιώ. Δεν υπάρχει συμφωνία για τη χρήση στην νομοθετική ε, πρωτοβουλία ε, κατ' εξουσιοδότηση ε, πράξεων, εκτελεστικών πράξεων. Δεν υπάρχει διοργανική συμφωνία και αυτό βράχει κυκλώνει και ε, μπλέκει τη νομοθετική ε, προσπάθεια. Έχω ίδια εμπειρία από την αναθεώρηση του κανονισμού 539 και το άλλο είναι η παραχάραξη του ευρώ. Αρκεί να κοιτάξει κανείς το Σέγγεν για να καταλάβει τι σημασία έχει αυτό που λέγω. Επιγόντως ε, θα πρέπει να υπάρξει διοργανική συμφωνία, αλλιώς δεν μπορούμε αποτελεσματικά να ανταποκριθούμε στο νομοθετικό μας έργο που μας αναλογεί. Ε, και είναι και συναπόφαση ε, από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Και ευχαριστώ και τελείωσα κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σκλοντ Μωράες. Δίδαγμα από πολλούς ομιλητές σήμερα ε, ως προς το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Στη χθεσινή συζήτηση, για παράδειγμα, που έγινε προφορική ερώτηση σε σχέση ε, με ε, την εγκατάσταση ετούντων ασύλων, μάθαμε πολύ γρήγορα ότι μετά τη διαδικασία στο δικαστήριο ε, εμφανίζεται μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας μια μεγάλη ανισορροπία μεταξύ ημών και ημών ε, του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και καλούμε ε, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει κάποια πράγματα επανειλημμένα. Είναι ο κοινός παρονομαστής πολλών βασικών θεμάτων που μας απασχολούν και πολλών προβλημάτων που έχουμε με την εφαρμογή. Και είναι πολλά τα κράτη-μέλη ε, που έχουν ε, θέματα με το άσυλο ε, έχουν ιδιαίτερο φόρτο ορισμένα ορισμένα άλλα κράτη είναι πρόθυμα να δεχθούν ανθρώπους που έχουν ζητήσει άσυλο σε άλλη χώρα, στη δική τους επικράτεια. Αυτά είναι μερικά από τα ζητήματα που μας απασχολούν. Δεν σημαίνει ότι δεν έχει επιτευχθεί πρόοδος όμως τα θύματα εγκληματικών ενεργειών, ε, διακίνησης ανθρώπων είναι άνθρωποι που ζητούν να ε, κάνουμε πρόοδο σε αυτούς τους τομείς και πρόοδο έχει γίνει. Αλλά ε, θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τις δυσκολίες με τρόπο αποτελεσματικό. Είπαμε για την παράνομη μετανάστευση. Μάλιστα, δεν είναι μόνο οι εποχιακοί εργαζόμενοι ε, αλλά και άλλοι έχουν πρόβλημα. Υπάρχουν προβλήματα με τα δικαιώματα των κατηγορουμένων δικονομικά και άλλα και θα πρέπει οπωσδήποτε να τα προωθήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος ε, Γιακολίνος Σαλβατόρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε έχουμε την αίσθηση ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης ε, τρία χρόνια μετά την έγκρισή του παραμένει ένα εργαλείο ανολοκλήρωτο. Αναφέρθηκε στις ε, παρεμβάσεις των ε, συναδέλφων και στην πρώτη παρέμβαση του Επιτρόπου κυρίου Μπόρκ ο οποίος τοποθετήθηκε υπέρ του Σέγκεν γιατί αναμφίβολα το Σέγκεν είναι ένα επίτευγμα του πολιτισμού ε, το οποίο έχει σχέση με, την, ε, με το πρόγραμμα Στοχόλμης. Είναι πολύ καλό το ότι υπάρχει συνεργασία των αστυνομικών δυνάμεων για να αντιμετωπίζετε καλύτερα το διασυνοριακό έγκλημα, το ξέπλυμα του βρώμικου χρήματος. Επίσης είναι το ότι υπάρχει και η προστασία των ανηλίκων. Αυτά είναι επιτεύγματα που καταγράφονται θετικά. Βεβαίως ε, υπάρχουν παρεμβάσεις ε, που δυστυχώς ε, δεν υλοποιήθηκαν ακόμα. Η δικαιοσύνη είναι ένα δικαίωμα, ένα δικαίωμα που πρέπει να εφαρμόζεται στην πράξη. Και αυτό το έχουμε προβλέψει και σε σχέση σχέση με τα σοφρονιστικά καταστήματα. Υπάρχουν και εκεί δικαιώματα. Ε, το πρόβλημα στα σοφρονιστικά καταστήματα είναι η συμφόρηση ε, και αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο ότι έρχονται πολίτες και από τρίτες χώρες. Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτα για να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση ε, στις ε, δημοσιονομικές ε, προοπτικές του 2014-2020 θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αυτό το πρόβλημα. Άρα δηλαδή υπάρχουν πολιτικές προτεραιότητες που είναι να αποδοθούν και πάλι ε, χρήματα αλλά και να αποδοθεί δικαιοσύνη έστω και με λιγότερα χρήματα. Νομίζω ότι επ' αυτού πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο συνάδελφος Βάιντεν Χόλτσερ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης που είναι ένα σημαντικό στοιχείο για την ασφάλεια, εσωτερική ασφάλεια της Ευρώπης δυστυχώς δεν έτυχε της αναγκαίας προσοχής ούτε στην ευρύτερη κοινή γνώμη από τους πολίτες ούτε από τους πολιτικά εμπλεκόμενους σε σχέση με αυτά τα μέτρα πολύ λίγο βρίσκονται στο προσκήνιο τα θεμελιώδη δικαιώματα και μόνο θυσιάζονται πολύ συχνά χάρη σε, σε μια προσχηματική ασφάλεια. Γι' αυτό θα πρέπει η αρχή της μη διακριτικής μεταχείρισης να διασφαλίζεται. Εξακολουθούμε να αναμένουμε την αξιολόγηση των νομικών διατάξεων σε σχέση με το Σέγγεν που στις 25 Νοεμβρίου είχε αποφασίσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2009. Είναι ένα ε, στοιχείο κλειδί αυτό για να καταπολεμηθούν αυτά τα θέματα. Υπάρχει και ένα μη νομοθετικό μέτρο που αναμένει ακόμα την έγκριση του Συμβουλίου σε σχέση με την ε, οδηγία. Αναμένουμε ακόμα να κατατεθούν. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Συνάδελφε, δέχεστε μία ερώτηση από τον κύριο Ερχάουζερ, παρακαλώ. Κύριε Ερχάουζερ, έχετε τον λόγο, παρακαλώ, για την ερώτηση. Αξιότιμε συνάδελφε Βάτεν Υπάρχει το απόφθεγμα ότι η ελευθερία θνίσκει με την ασφάλεια τούτου δεδομένου πιστεύετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δημιουργία ενός χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαίου βρήκε τη σωστή ισορροπία μεταξύ ασφάλειας αφενός και ελευθερίας αφετέρου. Τι λέτε, κύριε Βάιντεν Χόλτσερ, για αυτό το θέμα θα μπορούσε κανείς ε, επιμακρό να συζητήσει Πιστεύω ότι η ισορροπία αυτή τη στιγμή δεν έχει εξευρεθεί και ότι δυστυχώς όλο και περισσότερο κινούμεθα προς ε, μια κατεύθυνση μιας προσχηματικής δίθεν ασφάλειας ε, και απομένουν τα θέματα της ε, ελευθερίας σε πολλούς χώρους που εκκρεμούν. Περνάμε στη διαδικασία Catch the Eye. Η κυρία Μπασέσκου πρώτη, παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, σημαντικές πρόοδοι επετέχθησαν στην έγκριση του σχεδίου δράσης όσον αφορά το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις. Αναφέρομαι σε μία από τις πολιτικές προτεραιότητες αυτού του σχεδίου δράσης, την συνέχεια της διεύρυνσης του χώρου Σέγγεν δηλαδή, της επέκτασης του χώρου Σέγγεν. Ζητείται από το Συμβούλιο εκείνα τα κράτη τα οποία υλοποιούν τα αιτήματα του κεκτημένου του Σέγγεν να έχουν τη δυνατότητα να καταργήσουν τους ελέγχους στα σύνορα και η Ρουμανία και η Βουλγαρία υλοποιούν αυτά τα κριτήρια εδώ και πολύ χρονικό διάστημα και αυτό το ομολόγησαν και το επιβεβαίωσαν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αν επιθυμούμε την επιτυχία του προγράμματος της Στοχόλμης πρέπει αυτή η πολιτική προτεραιότητα διεύρυνσης του χώρου Σέγγεν να υλοποιηθεί και ελπίζω ότι μέχρι τα τέλη του 2013 θα επιτευχθεί αυτό. Πρόεδρο, σας ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω να ζητούν άλλοι τον λόγο. Και ο κύριος Επίτροπος μπορεί θα λάβει τον λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ πολύ και όλα τα μέλη τα οποία συμμετείχαν σε αυτή την ενδιαφέρουσα όντως συζήτηση. Για δέκα χρόνια ήμουν στη χώρα μου υπουργό ε, Εσωτερικών, οπότε αισθάνομαι αρκετά άνετα ε, με την συζήτηση αυτή. Κατανοώ τις ανησυχίες των μελών του Κοινοβουλίου και φυσικά ε, οι κυβερνήσεις κυβερνούν, έχουν αυτήν την υποχρέωση αλλά βεβαίως οι αποφάσεις τους θα πρέπει να ελέγχονται ενδελεχώς και αυτό κάνει ακριβώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ελέγχει ενδελεχώς ε, τι κάνουν τα κράτη-μέλη, πώς ε, υλοποιούν το κοινωτικό κεκτημένο και το κεκτημένο του Σέγγεν. Για να επανέλθω στον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησα την παρέμβασή μου, δηλαδή ότι η συνθήκη Σέγγεν είναι ένα επίτευγμα, ε, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθόλου ε, προβλήματα. Ο κύριος ε, Γκερέρο είπε ότι υπάρχουν δυσκολίες να πάει κανείς να ταξιδέψει από την Ευρώπη στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στο χώρο Σέγγεν. Ε, είχε τη δυνατότητα και την διακριτική ευχέρεια να μην προσυπογράψει την συνθήκη αυτή και επομένως μπορεί να ελέγχει τους όσους εισέρχονται στα σύνορά του. Καμιά φορά Ακούω και παράπονα από πολίτες ε, χωρών που ξέρω καλά, ε, όπου τους λένε ότι ακόμα και σε χώρες Σέγγεν δεν μπορούν να μπουν αν δεν έχουν θεωρημένο διαβατήριο ή καινούργιο διαβατήριο κτλ. Ε, υπάρχει και εκτιμένο το οποίο θα πρέπει να λειτουργεί σωστά και να μην υπάρχει καμία κατάχρηση ή καμία κακή χρήση της συνθήκη της συμφωνίας αυτής πίσω από τα παρασκήνια ε, και κρυφά να υψώνονται νέα τείχη και νέα προσκόμματα. Αυτό ισχύει και για όλη την φάση της υλοποίησης ε, του κεκτημένου του Σέγγεν. Ξέρω ότι κάποια μέλη αναφέρθηκαν ε, στο ένταλμα σύλληψης το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης, ότι δηλαδή μερικές φορές αδίκως χρησιμοποιείται κατά ορισμένων υπηκών, ενώ άλλοι καταγγέλουν ότι δεν χρησιμοποιείται αρκετά. Η ιδέα αυτού του Ευρωπαϊκού Εντάλματος βασίζεται στην υπόθεση ή στην αρχή μάλλον ότι προσωμιάζουν οι ε, ε, κανόνες μας για τον χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης δικαιοσύνης και επομένως αυτού του είδους το ένταλμα θα μπορούσε να αποτελεί έναν γρήγορο τρόπο ε, για τις απελάσεις γιατί βεβαίως υπάρχουν και οι συμφωνίες απέλασης βάσει και των αρχών του Συμβουλίου της Ευρώπης. Όμως εμείς πηγαίνουμε ένα βήμα παραπέρα. Εάν ε, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όπου εμπιστευόμαστε ένα τον άλλον ε, πολύ και όπου μοιάζουν και οι αρχές μας τότε μπορούμε να προχωρήσουμε ένα βήμα παραπέρα. Θυμάμαι τη μέρα που στο Ηνωμένο Βασίλειο υπήρξε έτσι μία ε, συζήτηση αντίθετη προς αυτό το ευρωπαϊκό ε, ένταλμα ε, σύλληψης Ε, συνέβη και το περιστατικό αυτού του ε, καθηγητού ο οποίος απήγαγε κατά κάποιο τρόπο ε, πήρε μία μαθήτριά του μαζί του στην Γαλλία και βεβαίως μέσω αυτής της διαδικασίας του Ευρωπαϊκού Εντάλματος μπόρεσε η Γαλλία να τον απελάσει με γρήγορες διαδικασίες. Ε, είναι μια απλουστευμένη μορφή απέλασης λοιπόν η οποία μπορεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις να βοηθήσει. Ε, αλλά φυσικά υπάρχουν πάντα περιθώρια έτσι ώστε να χρησιμοποιήσει κάποιος εσφαλμένα ή υπερβολικά αυτό το ε, εργαλείο. Όμως σε γενικές γραμμές, εάν λειτουργήσει, αν εφαρμοστεί σωστά και χρησιμοποιηθεί σωστά, τότε μπορεί να συμβάλλει στο χώρο ελευθερίας και δικαιοσύνης. Ευχαριστώ την ε, κυρία Ματζόνη από την Ιταλία για την δέσμευση, τη στράτευσή της ε, έτσι ώστε να γίνει η Ευρώπη ε, πιο, να αυξηθεί μάλλον η δημοκρατική λογοδοσία στην Ευρώπη έτσι ώστε να πιστούν και οι πλέον ευρωσκεπτικιστές για το καλό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω όμως ότι ε, το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμης και η θέσπιση του χώρου ελευθερίας ε, και δικαιοσύνης θα πρέπει να αξιολογηθεί όχι σε σχέση με το τι θα ήταν το ιδεώδες ή το τι θα θέλαμε όλοι, αλλά σε σχέση με το από ποιο σημείο ξεκινήσαμε. Πριν από μερικά χρόνια έπρεπε ε, οι υπουργοί να ξεκινήσουν από το μηδέν. Η κάθε χώρα μέλος, η Γερμανία και όλες οι άλλες χώρες, η κάθε μία ξεχωριστά, είχαν την δυνατότητα να ασκήσουν βέτο για κάθε απόφαση του χώρου ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σήμερα τα πράγματα έχουν αλλάξει υπάρχουν δύο συνομοθέτες ισότιμοι και το υπογραμμίζω αυτό, ισότιμοι που έχουν τα ίδια ακριβώς ε, δικαιώματα ε, και με ευχαριστεί κατά αυτή την έννοια η πολύ λογική προσέγγιση του κυρίου Μωράης ο οποίος είπε ότι η Κομισιόν έχει την ενεργητική κατά κάποιο τρόπο πλευρά ε, της ε, διαδικασίας. Ε, ήμουν 16 χρόνια μέλος της κυβέρνησης και πιστεύω ότι οι κυβερνήσεις τείνουν να είναι λίγο πιο συντηρητικές και λίγο πιο αργές στις αποφάσεις τους από ότι τα κοινοβούλια. Άλλωστε αυτό είναι και ο συμβιβασμός του να έχει κανείς αυτό που λέει ο πρόεδρος Μπαρόζο, μια ομοσπονδία που, που αποτελείται όμως από εθνικά κυρίαρχα κράτη. Δεν έχουμε γίνει πραγματική ομοσπονδία, αλλά από την άλλη πλευρά είμαστε κάτι πολύ περισσότερο από μια οργάνωση ε, κυριάρχων κρατών ε, και προχωρούμε προς μια πιο τέλεια ένωση. Απαντώ λοιπόν και στην ε, κυρία ε, Ματζόνη αν έχουμε μια πραγματική δύναμη ναι, έχουμε και έχουμε και μία δύναμη που είναι προωθητική. Απλώς ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο που θα επιθυμούσαμε και δεν αναφέρομαι σε ακαδημαϊκό επίπεδο αποφάσεων, αλλά αναφέρομαι στην ουσιαστική υλοποίηση. Υπάρχουν ε, και κάποια προσκόμματα τα οποία προκύπτουν κάθε τόσο και τα οποία είναι εθνικής ε, προέλευσης και τα οποία οπωσδήποτε θα πρέπει να λαμβάνονται άμεσα υπόψη έτσι ώστε να ξεπερνιούνται με άμεσες δράσεις. Στην ερώτηση πόση αλληλεγγύη υπάρχει όσον αφορά το θέμα της μετανάστευσης και βεβαίως οι περιφερειακές ε, ε, χώρες ε, παραπονιούνται ότι δεν έχουν γίνει αρκετά όσον αφορά την ενδοευρωπαϊκή μεταφορά ή ε, μετακίνηση μάλλον προστατευομένων ε, μελών και ότι η πίεση στην ε, περιφέρεια είναι πάρα πολύ μεγάλη όσον αφορά τους ετούντες άσυλο και τους πρόσφυγες. Κοιτάξτε, η, αλληλεγγύη συγγνώμη, δεν επιβάλλεται ε, ξέρετε ότι βεβαίως ε, απορρέει και από κάποιες υποχρεώσεις, αλλά παρόλα αυτά δεν μπορεί κανείς ε, να επιβάλλει ολοκληρωτικά ένα σύστημα μοιράσματος του άχθους. Αυτό το μοίρασμα του άχθους, αυτή η κατανομή η δίκαια θα πρέπει να αποφασιστεί από όλες τις χώρες. In Επομένως είναι θέμα αλληλεγγύης, αλλά καταλαβαίνουμε ότι αυτή η αλληλεγγύη δεν έχει προωθηθεί όσο θα έπρεπε από τα κράτη-μέλη. Θα πρέπει αυτό να ληφθεί υπόψη από όλα τα κράτη-μέλη ε, και να καταλάβουν όλοι ότι το πρόβλημα είναι πανευρωπαϊκό και επομένως θα πρέπει να πάρουν όλοι τις σχετικές αποφάσεις. Κοιτάξτε, θα ήθελα ε, να ε, συμφωνήσω με τον κύριο Γεύκα ότι ε, η κατάρτιση του προσωπικού της δικαιοσύνης ε, των δικαστικών είναι ε, κάτι πάρα πολύ σημαντικό και κατά αυτήν την έννοια η Κομισιόν θα εξακολουθήσει να στηρίζει τέτοιου είδους δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης γιατί με αυτόν τον τρόπο η νομοθεσία που έχει αποφασιστεί στο Στρασβούργο ή στις Βρυξέλλες δεν θα παραμείνει κενό γράμμα. Για το Σέγγεν έχω ήδη απαντήσει ερωτήματα. Όσον αφορά τώρα ε, μια άλλη ερώτηση ε, του κυρίου έρεν Χόζερ ε, πρέπει να σας πω ότι έχουμε δύο στόχους πρώτον να ε, κάνουμε την ε, Europol πιο, ε, πιο, αποτελεσματική και δεύτερον να αυξήσουμε την... τον έλεγχο του Κοινοβουλίου επί των δράσεων της Europol. Και ξέρετε ότι η παρέμβαση του Κοινοβουλίου είναι σημαντική για πολλά στοιχεία της νομοθεσίας ε, γιατί έχουν συζητηθεί πολλά πράγματα, έχουν επιτευχθεί πολλές ε, ε, συμβιβαστικές λύσεις και επομένως κανείς δεν πρέπει να αγνοεί τον άλλον, αλλά οι δύο συνομοθέτες σε συνέργεια αγαστή να μπορέσουν να βρουν αυτό το οποίο καλύτερα θα υπηρετήσει το συμφέρον της Ευρώπης. Σας ευχαριστούμε θερμά. Παρακαλώ, Ευχαριστώ πολύ. Αξιότιμα μέλη. <clears throat> Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μου δίνετε να έχουμε αυτόν τον διάλογο, τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ χρήσιμη για το πρόγραμμα της Στοκχόλμης. Όπως είπα εισαγωγικά, το πρόγραμμα αυτό καθεαυτό είναι ευρύτατο και περιεκτικό, συνολικό και περιλαμβάνει το άσυλο, τη μετανάστευση, την εσωτερική ασφάλεια, τις εξωτερικές σχέσεις και όπως τόνισαν πάρα πολλά μέλη, ε, το πρόγραμμα ε, και όλα τα στοιχεία ε, αυτού επηρεάζουν την ζωή των πολιτών με τον ένα ή άλλο τρόπο. όλες αυτές, όλα τα σκέλη της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων. Ε, συμφωνώ με τον φίλο μου Επίτροπο Μπόργ, διότι νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα benchmark, ένα σημείο αναφοράς αξιολογώντας από πού προήλθαμε. Βεβαίως όλοι ε, θέλουμε ε, το βέλτιστο αποτέλεσμα, ουτοπία ίσως, αλλά νομίζω ότι αξιολογώντας το πρόγραμμα ε, ε, που, έχει, που είναι πολύπλευρο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε διανύσει πάρα πολύ δρόμο. Θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικά από τα θέματα τα οποία τέθηκαν ειδικά από μέλη, ο κύριος Μπίλκερ, ε, και ο κύριος Κασίνη έχουν ε, διαρωτηθεί για τις πρακτικές, τα πρακτικά πλεονεκτήματα και τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί. Βεβαίως ο κατάλογος είναι μακρύς, αλλά νομίζω ότι τα αποτελέσματα που έχουν ε, επιτευχθεί νομίζω αποδεικνύονται από όλα τα νομοθετήματα στον το με αυτό εσωτερικών υποθέσεων νομοθετήματα που θα εξασφαλίσουν ε, την ασφάλεια σε κάθε άποψη της ζωής των πολιτών. Ο κ. Γκερέρο Σαλόμ ανέφερε την ανάγκη να εστιαστούμε σε αξίες και όταν μιλούμε για αξίες πρόκειται για τις ευρωπαϊκές αξίες που βρίσκονται στο επίκεντρο, που είναι ο πυρήνας του προγράμματος της Στοκχόλμης. Αναφέρθηκε ε, το θέμα της ε, μετεγκατάστασης, ε, όπως ξέρετε. Ένα πρόγραμμα υιοθετήθηκε τόσο από το Κοινοβούλιο όσο από το Συμβούλιο τον Μάρτιο πέρσι, ούτως ώστε να υπάρξει αντίδραση συντονισμένη σε αυτούς που απαιτούν, που ζητούν προστασία. Και η προστασία δίδεται ο κύριος Κέρκολ μίλησε για την πρόκληση ε, των ασυνόδευτων ανηλίκων. Πρόκειται και εδώ ε, για ένα θέμα που μας ανησυχεί, που μας απασχολεί, που απαιτεί την προσοχή μας. Τον Μάιο του 2010 η Κομισιόν παρουσίασε ένα πρόγραμμα δράσης ε, για την περίοδο 2010-2014 και η εφαρμογή αυτού του σχεδίου δράσης ε, αναφέρθηκε το Σεπτέμβριο ούτω ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα εξακολουθήσουμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά αυτόν ε, ε, την πρόκληση. Ο κ. Παπανόπουλου μίλησε για την νομοθετική διαδικασία μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Πιστεύω ότι η διαδικασία βελτιώθηκε σημαντικά με την διαδικασία της συναπόφασης και επίσης ο Επίτροπος τόνισε το σημείο αυτό. Νομίζω ότι η πλήρης δέσμευση του Κοινοβουλίου βελτιώνει τα πράγματα και ε, μας κρατά εμάς την Κομισιόν και το Συμβούλιο σε επαγρύπνηση. Νομίζω ότι αυτό είναι μεγάλη βελτίωση. Βεβαίως υπάρχει ακόμα πολλή εργασία που πρέπει να γίνει σχετικά με τις σχέσεις, τη συνεργασία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Αυτό απαιτεί βελτίωση αυτό βεβαίω ε, δεν υπάρχει μόνο στον τομέα της δικαιοσύνης και των εσωτερικών υποθέσεων, αλλά μέλη μίλησαν για την στρατηγική ε, διαχείρισης βεβαίως έχουμε ανταλλαγή μοντέλων ε, μια έκθεση δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο και θα πρέπει να κάνουμε έναν απολογισμό πώς ανταλλάσσονται διασυνοριακά οι πληροφορίες σήμερα ε, οι διαπιστώσεις της Κομισιόν εξετάζονται προσεκτικά για την ώρα από το Συμβούλιο. Και θα κάνουμε αναφορά. Ο κύριος Δίας Δημέρα ανέφερε ε, την οδηγία σχετικά με την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων ε, και αναφέρθηκε στην έλλειψη προόδου σχετικά με το θέμα αυτό. Ε, με χαρά μπορώ να πω ότι το πρώτο, πρώτος τριμερής διάλογος θα λάβει χώρο στις 28 Μαΐου ε, ακολουθώντας την Επιτροπή ΛΥΜΠΕ νομίζω ότι θα υπάρξει πρόοδος και ότι θα δείτε, θα δείτε ότι έχουμε εργαστεί σκληρά ε, για να έχουμε κάποια πρόοδο σχετικά με αυτήν την άποψη και άλλες απόψεις του προγράμματος της Στοχόλμης. Το πρόγραμμα αυτό καθε αυτό εξασφαλίζει ότι θέματα που θέλουν περαιτέρω ανάπτυξη και περαιτέρω προστασία, συνεχιζόμενη προστασία, να βρίσκονται στο επίκεντρο της προσοχής μας και αυτό είναι το πλεονέκτημα της προγράμματος της Στοκχόλμης ότι το θέμα παραμένει και διότι πρέπει να γίνουν βελτιώσεις και μεταρρυθμίσεις. Βεβαίως εξασφαλίσαμε τη συνέχεια ε, σε διάφορες προεδρίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, είναι, υπάρχει συνεργασία με το Κοινοβούλιο, ε, την Κομισιό, κατά τη διάρκεια των προεδριών που διαδέχονται η μία την άλλη. Αυτό είναι ευεργετικό. Ο τομέας της ελευθερίας, της ασφάλειας και της δικαιοσύνης για τον οποίο εργαστήκαμε τόσο σκληρά και να προστατεύσουμε έχει επηρεαστεί από τα διάφορα στοιχεία του προγράμματος. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω εν κατακλείδη ότι για την υπόλοιπη περίοδο και διάρκεια της Ιρλανδικής Προεδρίας θα εξακολουθήσουμε, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε πάρα πολύ σκληρά για να επιτύχουμε ε, πρόοδο στα πλαίσια του προγράμματος της Στοχόλμης και ε, ε, θα είμαι ευτυχής να έχουμε συνεχιζόμενη συνεργασία για να μπορέσουμε να συμβάλλουμε σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που αξίζουν νομίζω οι πολίτες μας. Πλησιάζει ίσως το τέλος της Ιρλανδικής Προεδρίας, το πλεονέκτημα του να έχει κανεί ένα πρόγραμμα όπω το πρόγραμμα της ε, Στοκχόλμη μας βάζει να εργαζόμαστε μέχρι την ε, τελευταία στιγμή και θα εργαστούμε για να ε, συνεχίσουμε ε, εποφελούμενοι από την όθηση που έχουμε ε, και από την συνεργασία του Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ και πάλι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ευκαιρία που μας δίνετε να συμμετάσχουμε σε αυτή τη συζήτηση. Σας ευχαριστούμε κυρία Προεδρεύουσα του Συμβουλίου. Σας ευχαριστούμε εμείς εσάς για το ότι όλη την ημέρα σήμερα παρακολουθήσατε τις εργασίες μας από πλευράς της Προεδρίας του Συμβουλίου ε, θέσατε πολύ ψηλά τη σημαία του Συμβουλίου. Ολοκληρώνεται αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερησίας διάταξης. Δήλωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση του θέματος του φόρου κληρονομιάς ε, όσον αφορά τον κανονισμό μετά την έγκριση του κανονισμού από πλευράς της Επιτροπής